Καλησπέρα σας. Το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι όπως πάντα η έγκριση της ημερησία διάταξη. Το σημείο 4, δηλαδή ψηφοφορία για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, θα μετακινηθεί και θα μπει μετά το σημείο 8. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη σε σχέση με τις ανακοινώσεις του Προέδρου. Έχω ένα σημείο. Πέρα από το μήνυμα ότι οι αποφάσεις των συντονιστών της 22ης Ιανουαρίου μπορούν να βρεθούν στο φάκελο της συνεδρίασης και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, επίσης θεωρείται ότι εγκρίνονται. Τώρα, η ενημέρωση που θέλω να σας δώσω είναι η εξής. Θέλω να σας ενημερώσω ότι έχουμε έναν αριθμό νέων ενημερωτικών σημειωμάτων διαθέσιμων ε, για το ε, επίμαχο θέμα των ε, καθαρών υπολείπων και για το πώς θα μετρηθούν τα ωφέλη του, ε, ναι, της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και του προϋπολογισμού. Αυτά τα έγγραφα έχουν παραχθεί από εξωτερικού συμβελμένους μετά απόφαση των συντονιστών. Η κυρία Αρμόν ήταν αρμόδια για τη σύμβαση αυτή. Τα σημειώματα εξετάζουν τη λειτουργία, το σκοπό, την ιστορία και τις ελλείψεις των διάφορων δικτών ιδίως σε ό,τι αφορά τα καθαρά λειτουργικά υπόλοιπα, τα οποία φυσικά βρίσκονται στο επίκεντρο της αιώνιας συζήτησης για τη δίκαιη επιστροφή. Φυσικά αυτό είναι ένα ιδιαίτερα επίκαιρο θέμα στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης συζήτησης για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ίσως ε, σε μια επόμενη συνεδρίαση να θέσουμε αυτό το θέμα στην ημερησία διάταξη με παρουσίαση των εγγράφων από τους συντάκτες τους και φυσικά θα έχουμε και την ανταλλαγή απόψεων που απαιτείται. Εν τω μεταξύ τα έγγραφα αυτά ήδη είναι διαθέσιμα δημοσίως και καλείται να τα λάβετε υπόψη και υπάρχουν στην αίθουσα και έντυπες εκδοχές των κειμένων. Κύριε Κέλλερ, ευχαριστώ. Είναι μεταφρασμένα τα έγγραφα αυτά, αυτά τα σημείωματα. Πρέπει να το ελέγξω, λέει ο Πρόεδρος. Όχι, όχι προς στιγμή. Θα δούμε αν ε, μπορέσουμε να τα μεταφράσουμε. Φαντάζομαι ενδιαφέρεστε για τη γαλλική εκδοχή. Είναι σημαντικά σημειώματα, επομένω ε, είναι καλύτερο για τον καθένα να μπορεί να εργαστεί στη γλώσσα του. Δεν ε, είμαι κατά να υπάρχουν και άλλες εκδοχές, γερμανική, σουδική, πολωνική, ουγγρική. Η πολωνική θα πρέπει να είναι προτεραιότητα είναι πολύ μικρός ο προπολογισμό. Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι ενδιαφέροντα τα έγγραφα αυτά. Ε, Επομένω, για την ε, συζήτηση του προπολογισμό που δεν έχει τελειώσει, είναι καλό να τα έχουμε. Θα το ελέγξουμε όμω πριν σα ε, δώσουμε υποσχέσει. Σχόλιο εκτό μικροφώνου. Let's, let's check before we... Να το ελέγξουμε πριν να αρχίσω να υπόσχομαι πράγματα που δεν μπορώ να τηρήσω. Σημείο 3 έγκριση των πρακτικών, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, επίσης θεωρείται ότι εγκρίνονται. So, we move to point five. Πάμε στο σημείο 5, το πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή τη Συμφωνία Σύμπραξη στον τομέα αλλία μεταξύ Δημοκρατία Ενεγάλη και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρουσιάστηκε και συζητήθηκε ο φάκελο αυτό στη συνάντησή μα στι 22 Ιανουαρίου. Να υπενθυμίσω ότι πρόκειται για διαδικασία συνένεση. Επομένω, ψηφίζουμε την γνωμοδότηση στο σύνολό τη. Πριν να περάσουμε σε ηλεκτρονική ψηφοφορία, να δούμε αν λειτουργούν τα μηχανήματα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πρόκειται για δοκιμαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε ό,τι θέλετε. Vote closed. Λήξη. 30 ψηφίσαντες. Εντάξει. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε λοιπόν την ελευτική σύμπραξη. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 26 υπέρ, 2 κατά και 2 εποχές. Ευχαριστώ. Σημείο 6 της ημερησίας διάταξης. Ε, έχουμε παράταση του πρωτοκόλλου για τον καθορισμό αληθικών δυνατήτων και χρηματική απαρχή που προβλέπουν τη Συμφωνία Σύμπραξη στον τομέα τη Ελία μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τη Ισλαμική Δημοκρατία τη Μαυριτανία, το οποίο λήγει στι 15 Νοεμβρίου 19, έληξε μάλλον στις 15 Νοεμβρίου 2019. Επίσης, συζητήθηκε στις 22 Νοεμβρίου στη συνεδρίασή μας και πάλι έχουμε εδώ διαδικασία συνένεση. Ψηφίζουμε λοιπόν το κείμενο στο σύνολό του. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Λήξη. Εγκρίνεται. 26 υπέρ, 3 κατά και μία αποχή. Πάμε στις μεταφορές, τμήμα 3, δεν ε, έχουν ληφθεί αιτήσει. Ε, σημείο 8, άλλα τμήματα για τις μεταφορές, κυρία Γουαρτία Σαμπάλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχουμε δύο σημεία επιτάπητος. Το ένα έχει να κάνει με τις 89 θέσεις ε, που έχουμε συζητήσει πολλάκις ε, σε αυτή την Επιτροπή και διαπραγματευτήκαμε κυρίως με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τη δίκηση του Κοινοβουλίου. Πρόκειται για μια μεταφορά θέσεων μεταξύ των ομάδων και της δίκησης προκειμένου όσοι μπορούν να επιλέξουν αυτή την ε, πασαρέλα μπορούν να κάνουν ε, τις πρακτικές και την εξέταση. Δεν ε, έχει δημοσιονομική επίπτωση. Απλώς ήθελα να σας ενημερώσω ότι η διοίκηση ζήτησε τη δημιουργία αυτών των 89 θέσεων και τη σχετική μεταφορά να αναφερθώ και στις μεταφορές για την Επιτροπή των Περιφερειών. Η Επιτροπή των Περιφερειών μας κάνει μία πρόταση, μία αίτηση μεταφοράς 255.000 ευρώ και μειώνονται οι μισθοί ενώ αυξάνονται ο προπολογισμό για τι δραστηριότητε που αφορούν την ενημέρωση των πολιτικών ομάδων. Μιλάμε μόνο για 255.000 ευρώ. Συνάδει με όσα ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν μιλήσαμε για τον προπολογισμό του 2020 για την Επιτροπή των Περιφερειών. Ζητήσαμε αύξηση αυτή τη γραμμή του προπολογισμού για να έχουμε περισσότερες δραστηριότητες στον τομέα της επικοινωνίας, όμως ήταν αδύνατο να πετύχουμε αυτό το κονδύλι και τώρα μας προτείνει μία μικρή διόρθωση, η Επιτροπή των Περιφερειών, ε, από το τμήμα των μισθών και σκεφτούμε το ποσό, είναι πολύ μικρό το 255.000, αλλά θα μπορούσε αυτό το ποσό να συνεισφέρει σημαντικά στο θέμα της πολιτικής επικοινωνίας των ομάδων της Επιτροπής των Περιφερειών. Ζητώ λοιπόν την υποστήριξη αυτής της Επιτροπής, γιατί όπως σας είπα συνάδει με τα όσα είχαμε προτείνει για τον προπολογισμό του 2020. Ευχαριστώ. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις... Όχι. Τότε θεωρούμε ότι εγκρίνεται η μεταφορά αυτή. Okay. Εντάξει. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Και το περνάμε λοιπόν στο σημείο 4, το οποίο το έχουμε αφήσει. Όπως σας είπα και στην αρχή. Αλλάξαμε τη σειρά δηλαδή. Το σχέδιο γνωμοδότηση το οποίο παρουσιάστηκε και συζητήθηκε στην συνάντηση στις 22 Ιανουαρίου Ας ψηφίσουμε με ονομαστική κλίση. Τροπολογία 1. Διανατάσταση χειρό. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Έγκρινεται. Τροπολογία 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβεβαστική 3 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 23 β. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εδώ θα χρειαστεί έλεγχος. 23 Β παρακαλώ. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται. Για την 10 υπέρ ψήφι και 19 κατά. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Επαλήθευση. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 24, παρακαλώ. Έναξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. Και περνάμε τώρα στη συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Δεν σηκώσετε καλά τα χέρια σας. Συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 10. Υπέρ. Κατά. Εδώ θα χρειαστεί έλεγχο πάλι. Έναρξη ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Και έτσι περνάμε στην τροπολογία 57α. Υπέρ. Κατά. Εδώ θα χρειαστεί πάλι έλεγχος. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 57 β. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 33 αποσύρεται. Συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η ε, συμβαστική 7, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 9, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. Η... Συγγνώμη, λέει η πρόεδρος, ε, ψηφίσουμε ακόμα την 65. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 66. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 67. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 68. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το σύνολο της γνωμοδότησης τώρα, όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική κλίση, έναρξη παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται με 26 ψήφου υπέρ, 2 κατά και 3 αποχέ. Και συγχαρητήρια στον εισηγητή. Sorry? Madame Marquez, Madame Marquez has the floor, please. Merci, Président. Η κυρία Μαρκές, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους και οδησίες για τη δουλειά τους, για τη δέσμευση που ανέλαβαν, για την σύνταξη αυτής της γνωμοδότησης ίδιας πρωτοβουλίας που κινητοποίησε πολλά μέλη και γι' αυτό συνεισέφεραν στη διαμόρφωσή της. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους θερμά. Πάμε στο σημείο 9 της ημερησίας διάταξης και το 10 ανταλλαγή απόψεων, building policies, η πολιτική για τα κτίρια, δεν ε, έχουμε λάβει κάτι. Άρα φτάνουμε στο σημείο 11. Να δούμε αν ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ο Γενικός Γραμματέας είναι παρόντες. Uh, Πέντε λεπτά διάλειμμα παρακαλώ, πριν έρθουν οι προσκεκλημένοι μας.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 Uh, Καλησπέρα και πάλι. Συνεχίζουμε την εξέταση της ημερήσιας διάταξής μας. Καλωσορίζουμε τον κύριο Βέλε, το Γενικό Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Σίλβερ Περέιρα, τον Αντιπρόεδρο. Η διαδικασία για τη σύνταξη του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ξεκινά το Φεβρουάριο. Οπότε και ο Γενικός Γραμματέας, τον οποίο έχουμε σήμερα μαζί μας, καταλήγει σε μια πρόταση καθορίζοντας τις προτεραιότητες και τους πόρους για την επόμενη χρονιά. Ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Βέλε, παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα το σχέδιο προϋπολογισμού στο Προεδρείο, που χρησιμοποιείται ως βάση για την υιοθέτηση των πρώτων προβλέψεων και εκτιμήσεων για ε, την κατάρτιση ενός προσχεδίου προϋπολογισμού, το οποίο υποβάλλεται στη δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Προσκαλέσαμε λοιπόν τον κύριο Βέλε, τον κύριο Περέιρα, για να προβούμε με αυτούς σε μια ε, βραχή ανταλλαγή απόψεων για τις προβλεπόμενες δαπάνες, αλλά και ε, έσοδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την οικονομική χρήση 2020-2021. Για να ολοκληρώσουμε τη χορογραφία μας να ζητήσω από τον κύριο Βέλε να πάρει το λόγο για 10 λεπτά περίπου και μετά να δώσω το λόγο στον κύριο Περέιρα για άλλα 10 λεπτά για να μας κάνει την παρουσίαση του προσχεδίου για τις προκαταρκτικές ε, ε, προβλέψεις εσόδων και δαπανών για την οικονομική χρήση 2020-2021. Ο κύριος Βέλε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. για την διαδικασία για το 2021. Νομίζω ότι καλό είναι ευθύ εξ αρχή ε, να σας υπενθυμίσουμε το χρονοδιάγραμμα την, Δευτέρα, την τελευταία Δευτέρα, την προηγούμενη Δευτέρα, όπως είπατε, έκανα την παρουσίαση αυτή στο Προεδρείο και σήμερα έχουμε τη δυνατότητα για πρώτη φορά να κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων σε ό,τι αφορά το Προεδρείο στις 19 Μαρτίου θα εγκρίνει την πρόταση και θα δώσει εντολή για την διαπραγμάτευση με την Επιτροπή προπολογισμού και στη συνέχεια θα έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε τις ε, διαπραγματεύσεις και αν όλα πάνε καλά στις, 13, στις 30 Μαρτίου θα μπορέσουμε να εγκρίνουμε το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων και στο Προεδρείο και στην Επιτροπή Προπολογισμού και στη συνέχεια θα ακολουθήσει και στην Ολομελία διαδικασία ε, με συνέχιση δυνάμει τον ε, Οκτώβριο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κρατά ε, κατά παράδοση 20% των διοικητικών εξόδων όλων των θεσμικών οργάνων. Παραδοσιακά, εδώ και πολλά πολλά χρόνια, λοιπόν, εδώ και δεκαετίε, το 20% πάει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στην προηγούμενη θητεία τώρα, το Κοινοβούλιο αποφάσισε να μην εξαντλήσει το πλαίσιο αυτό. Είχαμε το κεφάλαιο 5, το οποίο αυξήθηκε κατά μέσο όρο με πάνω από το 4% αλλά κατά κανόνα οι αυξήσει στο προϋπολογισμό του ευρωπαϊκού προπολογισμού ήταν 2, ε, κάτι, 3, κάτι. Άρα δημιουργήσαμε μεγάλο περιθώριο και είμαστε κάτω από το 20% αυτό το οποίο παραδοσιακά όπως σας είπα χρησιμοποιεί το Κοινοβούλιο. Αυτό τι σημαίνει ότι με μια ενδεχόμενη περικοπή στο νέο κεφάλαιο 7 είναι πολύ πιθανό και για το 2021 να μην υπερβούμε αυτό το 20%. Φυσικά, ο προϋπολογισμός ε, αφορά αριθμητικά στοιχεία, αλλά στην ουσία πίσω από τους αριθμούς ε, κρύβονται προγράμματα και έργα που βγάζουν νόημα, άρα θα πρέπει πάντα να εξηγούμε τι ακριβώς θέλουμε να πετύχουμε. Και γι' αυτό λοιπόν στο έγγραφο θα βρείτε μία σύντομη επισκόπηση σε ό,τι αφορά τα βασικά έργα και προγράμματα από την προηγούμενη θητεία. Τι δημιουργήσαμε, τι καινούριο δημιουργήσαμε με τα κονδύλια του προπολογισμού σε ό,τι αφορά και τις ε, διαβουλευτές μεταξύ Προεδρείου και Επιτροπής Προπολογισμού. Μία επιστημονική υπηρεσία. Ε, λοιπόν, δημιουργήσαμε και πολλές ε, θέσεις προήλθαν από άλλες υπηρεσίες οι οποίες έγιναν μετά από ανακατανομή στις Βρυξέλλες πλέον έχουμε την εξή κατάσταση. Ο κάθε Ευρωβουλευτή, πέρα από το δικό του γραφείο, έχει άλλα δύο γραφεία για του βοηθού του. Αυτό δεν ήταν έτσι στην προηγούμενη θητεία, στην αρχή τη προηγούμενη θητεία. Για πρώτη φορά λοιπόν στο Στρασβούργο πλέον έχουμε και ένα επιπρόσθετο γραφείο για τους βοηθούς γιατί υπήρχε μόνο ένα γραφείο παλιότερα το οποίο έπρεπε να το μοιραστεί ο Ευρωβουλευτής με το βοηθό από τη θητεία λοιπόν αυτή για πρώτη φορά έχουμε αυτό το ένα συν ένα, ε, τη ρύθμιση αυτή για τα γραφεία. Επενδύσαμε επίσης στον τομέα της ασφάλειας, κυρίως σε ό,τι αφορά τις εισόδους μετά τη δυσάρεστη εμπειρία που 200 Κούρδοι είχαν μπει από την είσοδο, διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρχε επαρκής ασφάλεια. Επίσης, ε, έγινε εσωτερική κατανομή των υπηρεσιών για του οδηγού. Έχουμε ανοίξει επίση τον οίκο για την Ευρωπαϊκή Ιστορία, το σπίτι τη Ευρωπαϊκή Ιστορία, ε, το οποίο το 2019 είχε 200.000 επισκέπτε. Το σπίτι τη Ευρωπαϊκή Ιστορία 200.000, ε, το Παρλαμεντάριουμ 300.000 ε, επισκέπτες και αυτό σε σχέση και με άλλα θεσμικά όργανα φτάνουμε περίπου στο 1 εκατομμύριο επισκέπτες και είχαμε και μία, ε, κάναμε μία πολύ επιτυχή ε, προεκλογική εκστρατεία σε όλα τα κράτη-μέλη και είχαμε περίπου 10.000 ε, νέους που συμμετείχαν και επίσης στις Βρυξέλλες είχαμε τρία νέα. Ανοίξαμε τρία νέα κτίρια. Το κτίριο Μάρτενς, χίλιοι υπάλληλοι, και επίσης χίλιοι υπαλλήλοι και στο Στρασβούργο το Χάβελ επίσης που φιλοξενεί χίλιους υπαλλήλου. Το νέο Προεδρείο λοιπόν στην αρχή της θετίας του τον Οκτώβριο έκανε ε, μία διάσκεψη στο Μαζός ε, έξω από το Παρίσι σε ένα κτίριο το οποίο μας ανήκει και το οποίο χρησιμοποιούμε για κέντρο για συνεδριάσεις και συζήτησε διάφορες στρατηγικές αποφάσεις τις οποίες και στη συνέχεια τις επισημοποίησε μέσω αποφάσεων του Προεδρείου. Και αυτό έχει σημαντικέ επιπτώσεις για τον προπολογισμό καταρχά. Η ευρωπαϊκή εμπειρία σε ό,τι αφορά δηλαδή αυτή τη μικρή διοργάνωση βουλών στα κράτη-μέλη, στη Φιλανδία για παράδειγμα, στη Γερμανία, στη Δανία, στη Σλοβανία, αυτό το μινι parliamentarium. Θέλουμε να επεκταθεί σε όλα τα κράτη-μέλη στην τρέχουσα θητεία. Αυτό θα είναι ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα και σημαίνει ότι θα έχουμε 12 νέες τέτοιες εμπειρίες κοινοβουλευτικές στο πρώτο ήμιση και 9 στο δεύτερο ήμιση της θητείας. Ο στόχος είναι να μην χρειάζεται ο κάθε πολίτης να έρθει στις Βρυξέλλες, στο Στρασβούργο. Να πάμε εμείς εκεί που βρίσκονται οι πολίτες και από την ε, εμπειρία μας στην Φιλανδία είχαμε πολύ θετικέ ε, ε, θετικά πορίσματα. Πολλοί επισκέφθηκαν αυτή την ευρωπαϊκή εμπειρία. Και φυσικά θα πρέπει να μην επικεντρωθούμε μόνο στις πρωτεύουσε, γι' αυτό πρέπει να είναι κινητό αυτό το κοινοβούλιο, το παρλαμεντάριο. Επίσης το Προεδρείο κατά αποφάσισε τους στόχου για το Πράσινο Κοινοβούλιο να του υλοποιήσει πιο γρήγορα και να είναι πιο προφιλόδοξη από ό,τι ω τώρα. Επίση έλαβε μια απόφαση μέχρι το 2024 να υπάρχει ισότητα μεταξύ φίλων σε ό,τι αφορά του διευθυντέ στο Κοινοβούλιο 50-50. Γιατί είμαστε τώρα στην, στο 40%. Και επίσης επιβεβαιώσαμε τις στατικές εμπειρίε μας από τις ευρωεκλογέ, όπου είχαμε 8% μεγαλύτερη προσέλευση στις κάλπες, 8 ποσοστιαίες ομα, μόναδες, από 42% σε 50%. Δηλαδή 34 εκατομμύρια επιπλέον ε, εκλογή. Και θέλουμε λοιπόν να ενισχύσουμε το έργο μας αυτό. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειάζεται παρουσία και στις εξωτερικές υπηρεσίες στα κρατη Επίσης, η στρατηγική για τα κτίρια αποφασίστηκε ήδη στα τέλη της προηγούμενης θετίας. Μετά από την θέση σε λειτουργία του κτηρίου Κόλ και Μάρτενς, να μην δημιουργήσουμε, γιατί δεν χρειαζόμαστε νέες υποδομές για γραφεία στις Βρυξέλλες, αλλά θα θέσουμε νέες προτεραιότητες. Καταρχά αυτή την εμπειρία τη Ευρώπη στα κράτη-μέλη. Κατά δεύτερον, η δυνατότητα τριμερών διαλόγων και απαραίτητων υποδομών, γιατί δεν έχουμε σωστού χώρου για τριμερεί διαλόγου. Και όταν χτίστηκαν τα κτίρια αυτά δεν υπήρχαν καν οι τριμερείς διαλογοί. Θα πρέπει να δημιουργηθούν λοιπόν σχετικέ δομές. Και τρίτον, ανακοινήσει. Το Κοινοβούλιο μέσονομοθεσία έχει αποφασίσει κάθε χρόνο να ανακοινήσεται ένα 3% των ε, κτίριων που κατέχει. Αυτό το κριτήριο λοιπόν θα πρέπει να ισχύσει και για τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα αλλά και για το Κοινοβούλιο, Επίση, τα κτηριακά. Έχουμε διάφορα έργα τα οποία θα ολοκληρωθούν σύντομα. Για παράδειγμα, φέτο θα έχουμε το πρώτο ανατολικό τμήμα του κτηρίου Adenauer που θα ανοίξει για την πρώτη Γενική Διεύθυνση ΙΜΛΟ, η οποία είχε ήδη εγκατασταθεί. Για 3.000 υπαλλήλου, επίση για όλου του υπαλλήλου μα ε, στο Λουξεμβούργο, 70% ε, το δυτικό, η δυτική πτέρυγα είναι το 30% εκπροσωπεί 16,2 εκατομμύρια και δεν έχει ακόμα ετοιμαστεί στο Στρασβούργο τώρα. Έχουμε να ολοκληρώσουμε το κτίριο για την ασφάλεια. Ως τώρα είχαμε υπολογίσει 8 εκατομμύρια ευρώ κόστος προσωρινά. Στις Βρυξέλλες έχουμε το, το, δύο, το κτίριο Atrium, το οποίο θα φιλοξενήσει ένα νέο κέντρο για επισκέπτες. Και κυρίως στη φάση ε, ανακαίνησης θα έχουμε λοιπόν ε, ένα μεγάλο κέντρο επισκεπτών 2,4 εκατομμύρια ευρώ και το info, το κέντρο ενημέρωσης ε, θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2021. Έχουμε επίσης και άλλα projects σε ό,τι αφορά το IT, σε ό,τι αφορά το hardware. Έχουμε δύο πολύ σημαντικά προγράμματα. Καταρχάς την αντικατάσταση όλων των ε, υπολογιστών desktop με βρετικούς υπολογιστές μέχρι το 2024 γιατί οι βρετικοί υπολογιστέ ε, επιτρέπουν ε, και την ε, κινητή, τη μετακίνηση στην εργασία. Δεν χρειάζεται να είναι κανεί στο ίδιο γραφείο και αυτό δεν είναι ευελιξία για να μπορεί να εργάζεται από το σπίτι του αλλά και στο κοινοβούλιο. Για να υπάρχει αυτή η ισορροπία μεταξύ εργασιακού και επαγγελματικού και οικογενειακού βίου. Και είχαμε και επίσης διάφορες ε, συσκευές οι οποίες έχουν ήδη αντικατασταθεί. Θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2024. Επίσης θα χρειαστούμε πιο υψηλά πρότυπα σε ό,τι αφορά τα κέντρα δεδομένων, data center γιατί το τρέχον κέντρο δεδομένων έχει κατηγορηποίηση ΑΑ. Χρειαζόμαστε τετραπλό Α όμως για να πετύχουμε το επίπεδο ασφάλειας που θέλουμε. Εδώ θέλουμε λοιπόν νέους παρόχους, τους οποίους θα πρέπει να ζητήσουμε. Τελευταίο σημείο σε ό,τι αφορά αυτή τη γενική εισαγωγή, σε ό,τι αφορά τα θέματα προσωπικού. Έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα περικοπής του προσωπικού κάναμε περικοπή όχι 5% όπως ζητούταν, αλλά μεταξύ 6 και 7% γιατί είχαμε κάνει αποζημίωση σε ό,τι αφορά το προσωπικό των πολιτικών ομάδων με μια ιστορική δίκλυτα. Θα... Η μοναδική πρόταση που γίνεται εδώ είναι οι πολιτικές ομάδες να, κάνουν, να δώσουν παράταση για 89 θέσεις μέσω του προγράμματος Πασαρέλα. Σε ό,τι αφορά και την, για ε, ε, να διατηρήσουν μάλλον τους υπαλλήλου από τις πολιτικές ομάδες, αν το επιθυμούν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Αδίνω τώρα το λόγο στον κύριο Περέιρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον Γενικό Γραμματέα και όλους τους ε, συναδέλφους. Θα ήθελα να σας χαιρετήσω και ε, να πω το εξή. Θα είμαι πολύ σύντομος και δεν θα εξαντλήσω το χρόνο που δόθηκε γενναιόδωρα. Γιατί στο στάδιο που βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά την διαδικασία του προπολογισμού, εγώ θα ήθελα όλοι να κατανοήσουν ότι ήδη έχουμε μία προκαταρκτική πρόταση προπολογισμού για το επόμενο έτος, όμως αυτή δεν είναι ακόμη η πρόταση του Προεδρείου. Σύμφωνα με την ε, διαδικασία μας, ο Γενικός Γραμματέας παρουσιάζει μία προκαταρκτική πρόταση, γίνεται μία πρώτη συζήτηση, έγινε μία πρώτη συζήτηση σε επίπεδο Προεδρίου, όμως ε, το Προεδρείο υιοθετεί την πρόταση προϋπολογισμού ε, μόνο μετά τις 9 Μαρτίου, την επόμενη μέρα και την επόμενη 9 Μαρτίου δηλαδή, 9 Μαρτίου και θα ήθελα να αναφερθώ στην ανταλλαγή απόψεων που γίνεται εδώ στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και ακριβώς αυτό το σκοπό και παρουσία μου να υπάρξει δική μου συμμετοχή ε, στη συζήτηση προκειμένου οι ανησυχίες όλων των συναδέλφων να αντικατοπτριστούν στις συζητήσεις που θα έχουμε στο Προεδρείο σχετικά με την πρόταση προϋπολογισμού. Επομένως, η δική σας συνεισφορά είναι μεγίστης σημασίας για το Προεδρείο του Κοινοβουλίου. Λεγθέντος αυτού. Θα ήθελα να πω, έχοντας φυσικά υπόψη και την αρχική συζήτηση που κάναμε στο Προεδρείο, ότι η πρόταση που παρουσιάστηκε από το Γενικό Γραμματέα. Όσοι είναι γνωστό, ενέχει μία συνολική αύξηση του προϋπολογισμού της τάξης 3,5% και αυτή η διαφοροποίηση, αυτή καθ' αυτή, δεν είναι ούτε κάτι λίγο ούτε πολύ. Θα πρέπει να αξιολογήσουμε αυτή τη διαφοροποίηση του προπολογισμού σε σχέση με τις προτεραιότητες και με τις αναγκαιότητες για να δούμε αν ε, αυτή η αύξηση είναι παραπάνω από όσα χρειαζόμαστε ή δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μας. Και εγώ νομίζω ότι είναι ορθό να υπογραμμίσω καταρχήν, γιατί αυτό τον, προβληματισμό έκανε και το Προεδρείο ότι η πρόταση προπολογισμού συνάδει με προηγούμενες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και του Προεδρείου. Και επομένως θεσπίζει μία σειρά προτεραιοτήτων που φαίνεται να είναι προτεραιότητες που καλύπτουν τις δικές μας ανησυχίες. Στην πραγματικότητα, οι κύριες αυξήσεις που βλέπουμε σε αυτή την πρόταση προϋπολογισμού έχουν να κάνουν με τις συνθήκες εργασίας στο Κοινοβούλιο. Μιλάμε και για εξοπλισμό ε, και σε ό,τι αφορά εξοπλισμό σε έπιπλα αλλά και σε υπολογιστές. 10% κατόπιν ε, σε θέματα ε, μελετών και ενημέρωσης ε, προκειμένου να υποστηριχθεί το έργο των βουλευτών και των ομάδων τους της τάξης του 15%. Όμως εμείς θέλουμε να δούμε εδώ όχι μόνο τις μεταβολές αλλά και για το ποιου τομεί θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη δημοσιονομική προσπάθεια. Αυτές οι επενδύσεις που έχουν γίνει αποτελούν συνέπεια των προηγούμενων αποφάσεων. Έχουμε ουσιαστικές επενδύσεις σε ό,τι αφορά τα κτίρια και την ασφάλεια. Ήδη υπόθηκε αυτό. Κυρίως αναφέρθηκε το κτίριο Αντενάουρ στο Λουξεμβούργο αλλά και εδώ το κτίριο ΣΠΑΚ της Βρυξέλλες. Επίσης, είχαμε επενδύσεις πρόσθετες στον τομέα της ασφάλειας, που είναι απαραίτητες και πρέπει να δοθεί και μια υποστήριξη στην υποδοχή των επισκεπτών και στο Στρασβούργο αλλά και στις Βρυξέλλες. Δεύτερο σχόλιο. Να πω ότι υπάρχει μία ανησυχία για τον προϋπολογισμό του επόμενου χρόνου, δηλαδή θέλουμε να καλυφθεί το θέμα της ενημέρωσης και της επικοινωνίας. Είναι προφανές ότι αυτές οι επενδύσεις προκύπτουν από προηγούμενες αποφάσεις, ιδίως σε ό,τι αφορά την ε, διεύρυνση του προγράμματος Europa Experience. Επίσης, είχαμε και την ιδέα του κινούμενου βουλευτή και το θέμα της σημασίας ε, των εκστρατεών ε, για την ευρωπαϊκή εκπαίδευση. Είναι αυτό κάτι πολύ σημαντικό και εγώ θα έλεγα πολύ περισσότερο σήμερα με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ευρωπαϊκό σχέδιο. Και ένα τρίτο σχόλιο για να τονίσω τις επενδύσεις στο θέμα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Έχουμε ένα κονδύλι 11,3 εκατομμύρια ευρώ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Και φυσικά αυτή η πτυχή είναι όλα και πιο σημαντική στη δυναμική του Κοινοβουλίου. Εμείς μάλιστα κληθήκαμε από το σύστημα εσωτερικού λογιστικού ελέγχου και μας επεσήμεναν ε, τις ε, ευάλωτες πτυχές που υπάρχουν ακόμα και την αναγκαιότητα να ενισχύσουμε την ε, ικανότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο θέμα αυτό. Επομένως, έχουμε τα θέματα της ασφάλειας στον ε, κυβερνοχώρο, ε, το θέμα της επικοινωνίας, είναι πολιτικές προτεραιότητες αυτές που τις βλέπουμε να αντικατοπτρίζονται στον προϋπολογισμό και φαίνεται να συνάδουν με προηγούμενες συζητήσεις και ανησυχίες που είχαμε εκδηλώσει. Λοιπόν, για να κλείσω. Κάποιες ε, ανησυχίες που εκφράστηκαν στο Προεδρείο και θα θέλαμε να μεταφραστούν στην τελική εκδοχή του προπολογισμού και θα δούμε τώρα πώς αυτό θα καταστεί δυνατόν, είναι τα εξή. Καταρχήν, ενίσχυση της ικανότητάς μας σε ό,τι αφορά τη διερμηνία και τη μετάφραση και θα υποστηρίξουμε λοιπόν το έργο των διερμηνέων προκειμένου να καλύπτονται και απαιτήσει. Δεύτερον, εκφράστηκε η ανησυχία να επαληθεύσουμε σε ποιο βαθμό το κονδύλι για τους ε, κοινοβουλευτικούς βοηθούς μπορεί να λαμβάνει υπόψη τις αυξημένες ευθύνες που προκύπτουν ε, κατόπιν του Brexit και να υπάρχει μια ενίσχυση ε, και των ομάδων ε, των βουλευτών προκειμένου η βοηθή που υποστηρίζουν τους βουλευτές της Βρυξέλλες και στους τόπους εργασίας δηλαδή του Κοινοβουλίου να ενισχυθούν και να μπορέσουμε να βρούμε μια κατάλληλη λύση, πιο κατάλληλη λύση. Και τέλος, το θέμα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Γιατί, όπως είπα προλίγου, αυτό αποτελεί προτεραιότητα. Και πέρα από την δημοσιονομική προσπάθεια που προβλέπεται σε αυτή την πρόταση προϋπολογισμού, θα πρέπει να ελέγξουμε αν μπορούν να καλυφθούν οι απαιτήσει και οι ανάγκες. Αυτά τα σχόλια θέλω να κάνω εισαγωγικά για τη συζήτησή μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Thank you, uh, Mr. Ευχαριστώ τους κυρίους Βέλε και Περέιρα για τις εισαγωγικές τους παρατηρήσεις. Ξεκινά τώρα η συζήτηση. Να δώσω καταρχάς το λόγο στον κύριο Σαστέλ, τον εισηγητή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Γενική Γραμματέα, κύριε Αντιπρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πολύ διότι μας εξηγήσατε με πολλές λεπτομέρειες αυτό το προσχέδιο προϋπολογισμού για τις δαπάνες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την οικονομική χρήση 2020-2021. Παρουσιάζεται αυτό το προσχέδιο ως στραμμένο προς το μέλλον και προς την νεωτερικότητα. Απαριθμίσατε έξι τομείς προτεραιότητες και ζητάτε προϋπολογισμό 2 δις 110 εκατομμύρια εκατομμύρια ευρώ, κάτι το οποίο αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 3,52% συγκριτικά με τον προϋπολογισμό της προηγούμενης οικονομικής χρήσης 2019-2020, 72 εκατομμύρια αύξηση και 32 από αυτά σχετίζονται με υποχρεώσεις που προβλέπονται από το καταστατικό ή από συμβάσεις που έχει υπογράψει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι αυτονόητο ότι η Επιτροπή για τον Προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να αναλύσει με εμπεριστατωμένο τρόπο και με με αυστηρότητα τις προτάσεις σας εν ώψη και του μελλοντικού πλαισίου για το, ε, και του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και για να είναι, έχει αξιοπιστία σε σχέση με τα άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον οποίο τον προπολογισμό εμείς αναλύουμε και ψηφίζουμε. Με άλλα λόγια, είναι πολύ δύσκολο να ασκούμε κριτική στον προπολογισμό των άλλων όταν δεν έχουμε ασκήσει κριτική στον δικό μας προπολογισμό. Γι' αυτό και θα το πράξουμε. Οι φιλοδοξίε σας ε, ξεπερνούν ε, τα εσκαμένα ε, είναι ε, παραπάνω από την απλή αύξηση λόγω αριθμοποίηση και τίποτα άλλο. Θα πρέπει όλα αυτά λοιπόν να τα αναλύσουμε πάνω σε ποια κριτήρια βασίζονται και το καθεξής. Βεβαίως σημείωσα επισταμένους του τομείς και τα σχέδια στα οποία θέλετε να δώσετε άμεση προτεραιότητα, π.χ. Ε, η επικοινωνία με το πολίτη, το σχέδιο για το κτηριακό, το σχέδιο για την ασφάλεια. Υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα και έργα για την ασφάλεια, εσωτερική ανάληψη του θέματος της ασφάλειας Λουξεμβούργο, κύβερνο ασφάλεια, εξυγχρονισμό των υποδομών μας και ειδικά των υπηρεσιών διασκέψεων και συνεδρίων, ανάπτυξη των ε, τεχνολογιών πληροφορικής και ε, ε, αηφόρο ανάπτυξη και κοινοβούλιο και κινητικότητα. Είναι όλοι αυτοί οι τομεί στου οποίου αναφερθήκατε. Θα ήθελα να ξεκινήσω με το πρασίνισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αυτό το οποίο ανέφερα τελευταίο. Η κλιματική αλλαγή αποτελεί οριζόντια προτεραιότητα για όλε τι πολιτικέ μα ομάδε. Θα ήθελα να γίνει μια διαπίστωση τη κατάσταση, μια αναφορά για, για τα ενεργοβόρα κτίρια, για το η ενέργεια καταναλώνουν όλα τα κτίρια τα οποία χρησιμοποιεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχετε επισκεφθεί διάφορα κτίρια στα οποία στεγαζόμαστε και κύριε Γενική, Γραμματέα μιλήσατε για το κτίριο Wilfried Martens, το οποίο είναι υπόδειγμα για το θέμα αυτό και θα ήθελα να ξέρω τι συμβαίνει και με τα λοιπά κτίρια από πλευράς περιβαλλοντικών κανόνων και θα ήθελα να γνωρίζω ε, περισσότερο τι θα υλοποιήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ποιε δράσει θα εφαρμόσει για να ενθαρρύνει το προσωπικό του και εδώ στη Βρυξέλλες αλλά και στο Στρασβούργο για να μειώσει τη χρήση των ΙΟΤΑΧΗ και να δώσουν προτεραιότητα προτεραιότητα ε, στη χρήση ε, των δημοσίων μέσων ε, μεταφοράς, στη δημόσια συγκοινωνία να στραφούει το προσωπικό ή και στο ποδήλατο. Επίσης, ποια είναι η πολιτική που θα, έχετε, θα υιοθετήσετε για τη χρήση των υδάτινων πόρων και της ηλεκτρικής ενέργειας. Δεύτερη σειρά ερωτήσεων που έχει να κάνει με το κτηριακό είναι μια σειρά ερωτήσεων για την οποία έχετε εν μέρει απαντήσει. Μιλούμε για το μέλλον του κτηρίου PHS εδώ ΠΕΑΣΕΣ εδώ στι Βρυξέλλες για την ανακαίνιση του κτηρίου, τον εξυγχρονισμό του για τη βελτίωση των ε, υποδομών ε, για τι συνεδριάσεις. Άκουσα ότι υπάρχει ένα έγγραφο για την κτηριακή στρατηγική μετά το 2020-2021. Δεν μπόρεσα να το βρω. Δεν ξέρω αν έχετε αντίγραφο εδώ ε, αυτού του εγγράφου για να μπορέσω να του ρίξω μια ματιά. Σε γενικέ γραμμέ, σε σχέση με την πολιτική σα για το κτηριακό, επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σα την άποψή μου είναι πραγματικά περίπλοκο το ζήτημα. Ορισμένα μέλη της Επιτροπής μας ε, έχουν προβληματιστεί διότι δεν εξηγείται αρκετά ε, το θέμα της αποκομιδής σε σχέση και με το κτηριακό και πάντοτε το κάνετε αυτό στο τέλος της κάθε θητείας. Δηλαδή, στο τέλος της κάθε θητείας ε, πολύ γρήγορα κλείνονται τα θέματα του κτηριακού. Πιστεύω ότι πρέπει να είστε πιο παιδαγωγικοί να εκπαιδεύσετε τα μέλη περισσότερο, να καταλάβουμε καλύτερα πώς επενδύει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και εκτός στη Νέα Υόρκη, στη Τζακάρτα μεταξύ άλλων. Οι επενδύσεις του Κοινοβουλίου είναι σημαντικές. Θέλω να χαιρετήσω τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της παρενόχλησης των διακρίσεων με βάση το σεξουαλικό προσανατολισμό. Έχουμε νέες δομές ε, και για την καταπολέμηση της παρενόχλησης ε, σε ομοφιλοφίλους και νομίζω ότι υπάρχει μια τέτοια δομή και θέλουμε να μας πείτε για τα αποτελέσματα αυτής της δομής, αυτή η νέα διαδικασία αν έχει ωφέλη και ποια ήταν αυτά. Θέλω να σας μιλήσω για τη θαυμάσια εμπειρία που ήταν το European Youth Event. Οι προηγούμενες εκδόσεις πράγματι και αυτές είχαν στεφθεί με επιτυχία. Ε, για προφανείς λόγους εγώ θα ήθελα να γνωρίζω το εξής. Μήπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει μόνο να στέλνει προσκλήσεις απανταχού στην Ευρώπη για να συμμετάσχουν οι νέοι, αλλά και να καλύψει τα έξοδα μετάβασης και ταξιδίου των νέων αυτό. Ναι. Είναι θέμα ισότητας εναντί των νέων. Ορισμένοι δεν μπορούν να πληρώσουν οι το ταξίδι του, ούτε τη στέγασή του εδώ για να ταξιδέψουν μέχρι εδώ στι Βρυξέλλε και να επισκεφθούν τα θεσμικά όργανα. Καλό θα ήταν το Κοινοβούλιο να μπορέσει να καλύψει αυτά τα, τα έξοδα. Και θα ήθελα να σταθώ και στις συνέπειες του Brexit, στις οποίες αναφερθήκατε πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε. Στο κείμενο του Γενικού Γραμματέα διάβασα ότι οι οικονομίες, η εξοικονόμηση που ε, που αποκτήσαμε λόγω της αποχώρησης των Βρετανών βουλευτών απορροφήθηκε η εξοικονόμηση αυτή από το προϋπολισμό του 2020. Δεν καταλαβαίνω γιατί το 2021 αυξάνουμε σε σχέση με το 20 και το 2019 τα έξοδα μετάβασης και ταξιδίου των ευρωβουλευτών ενώ έχουμε λιγότερους ευρωβουλευτές και έφυγαν οι Βρετανοί και έχουμε λιγότερες έδρες στο σύνολο. Έχουμε τους βοηθούς 4.220 είναι η γραμμή του προϋπολογισμού, αυξάνεται η γραμμή αυτή το 2021 σε σχέση με το 20 και το 19 και πρέπει να τα εξηγήσετε αυτά. Αξίζουν εξήγηση, υπάρχω, ε, ε, πιστεύω, αν υπάρχει εξήγηση. Και τέλος. Μιλήσαμε για το θέμα των ε, προφορικών επεξηγήσεων ψήφου. Θέλω να χαιρετήσω την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν οι διερμηνείς αλλά και οι μεταφραστές στο γραπτό κείμενο. Κάνουν μια δύσκολη δουλειά σε δύσκολες συνθήκες. Θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξορθολογίζει ορισμένα πράγματα. Θα πρέπει, χρειάζεται πραγματικά η προφορική επεξήγηση ψήφου κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας, ενώ μπορεί κανείς να εκφράσει την άποψή του για το πώς ψήφισε με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους και να απευθυνθεί στην κοινή γνώμη. Την περασμένη χρονιά, κύριε Γενική Γραμματέα, μας εξηγήσατε και μας είπατε ότι οι προφορικές επεξηγήσεις οι, προσωρινές, οι ψήφου στην Ολομέλεια πέρσι μας είχατε πει ότι στοιχίζουν 900.000 ευρώ ε, και νομίζω ότι καλό θα ήταν να γίνει εξοικονόμηση γιατί πραγματικά πιστεύω ότι δεν τη χρειαζόμαστε. Την προφορική επεξήγηση ε, ψήφου. Περιμένω τις απαντήσεις σας λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Βίντσι παρακαλώ. Αξιότιμη κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Γενική Γραμματέα, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, παρέμβαση αυτή. Είμαι από του καινούργιου Ευρωβουλευτέ και προφανώ ε, μου λείπουν κάποιε πληροφορίε, αλλά φυσικά και είναι σημαντικό το τι κάνουμε με τα χρήματα των φορολογουμένων. Και αυτό φυσικά και στα εθνικά κοινοβούλια. Στην έκθεσή σα ε, μιλήσατε και επισημάνετε πόσο σημαντικό είναι να αισθάνονται ε, κοντά στην Ευρώπη οι πολίτε. και είπατε ότι θα έχουμε μια τετραετή προεκλογική εκστρατεία. Τι εμπειρίες έχετε από το παρελθόν, Πώ θα δημορφωθεί αυτή. επίση κάτι άλλο που με έκανε εντύπωση, ποια είναι η διαφορά μεταξύ τη εμπειρία Europe Experiences και του Parliamentarium, ε, του μίνι Parliamentarium. Υπάρχει κάποια διαφορά, είναι το ίδιο. Επίσης είχαμε το θέμα της Πράγας και της Στοκόλμης που είχαν μπει στο προϋπολογισμό. Έχουμε άλλες πόλεις τώρα αυτή τη φορά. Αυτό που οφείλεται στο θέμα της ασφάλειας της εισόδου του κτηρίου. Τα συνολικά έξοδα είναι 11,3 εκατομμύρια. Αυτό αναφέρεται. Χτες 6 εκατομμύρια είχαν μπει στο προϋπολογισμό και 8 τώρα. Εδώ δεν μου βγαίνει η πρόσταση σε ό,τι αφορά την ασφάλεια στο Λουξεμβούργο. 150 νέοι υπάλληλοι. Γιατί προσλαμβάνονται τώρα και γιατί δεν έχουμε μία εταιρεία ασφάλειας. Αυτό μου κάνει κάποια εντύπωση. Κοιτώντα επίσης την ιστοσελίδα της ΕΠΣΟ, αυτές ε, οι 150 θέσεις έχουν ε, προκηρυχθεί παρόλο που δεν έχει αποφασιστεί ο προϋπολογισμός ακόμα και για το Brexit. και για τη μείωση του αριθμού των ευρωβουλευτών θα έχουμε 46 λιγότερους ε, ευρωβουλευτές και 160 λιγότερους ε, αμα, βοηθούς. Εγώ θεωρώ ότι θα δυσκολευτούν να εξηγήσω στην εκλογική μου περιφέρεια ότι θα αυξηθούν τα έξοδα ταξιδίου παρόλα αυτά. Ευχαριστώ. Mr. Ευχαριστώ κύριε Ουζακοφς. Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Θα ήθελα να θέσω κάποιες ερωτήσεις για τους πρόσθετους πόρους, ε, γιατί βλέπουμε μια αύξηση να έχει σχεδιαστεί 3,5% και αυτό σημαίνει ότι έχουμε ε, ε, περίπου 40 εκατομμύρια που είναι ελεύθερη επιλογή για την πρόσθετη χρηματοδότηση. Μήπως θα μπορούσαμε να έχουμε ένα πίνακα για το πώς προτίθεστε να ξοδέψετε αυτά τα 40 εκατομμύρια θα ήταν ε, πολύ χρήσιμο για τους βουλευτές ε, να δουν αυτό το πίνακα, δηλαδή πώς ε, θα δαπανηθούν αυτό τα χρήματα και επίση αν μιλάμε για τα νούμερα στο προσχέδιο. Βλέπουμε στο 32 σε ό,τι αφορά την εμπειρογνωμοσύνη στην επικοινωνία έχουμε μία αύξηση 15,7%. Γιατί τόσο υψηλή η αύξηση Επίσης, ε, μιλάμε κυρίως για ανθρώπους που δουλεύουν ως βοηθούς. Ακούσαμε τα σχέδιά σας ε, για τους βοηθούς μετά τον Brexit. Μήπως μπορείτε να μας πείτε κάποιες λεπτομέρειες. Και το τελευταίο που σχετίζεται με το προπολογισμό και υπάρχουν ε, πολιτικοί λόγοι είναι το Europe Experience. Πιστεύω ότι είναι πολύ ωραίο που έχουμε τρεις ε, τέτοιε αντιπροσωπείες στη Γαλλία, Παρίσι, Στρασβούργο και στο Βασόξ, αλλά στη Βαλτική, παραδείγματο χάρη, στις τρεις χώρε τη Βαλτική που έχουμε ιδιαίτερα πολύ πλοκή ευρωπαϊκή εμπειρία, θα θέλαμε μια μέρα να δούμε κι εμείς κάτι τέτοιο και το χρειαζόμαστε. Έτσι λοιπόν ε, είναι και το θέμα της ανισορροπίας σε ό,τι αφορά τις δαπάνες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριος Μπουζελακές. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση. Εδώ είμαι από την ομάδα των Πρασίνων θέλουμε να κατανοήσουμε ουσιαστικά τα δύο αποτελέσματα του σημερινού προπολογισμού και τις αλλαγές στην πρότασή σας, το χάρη στο κόστος ε, της ενέργειας ε, που ευξάνεται. Θέλετε να αυξήσετε σε όγκο ή σε τιμές ε, και ναι, θα ήθελα να καταλάβω λίγο καλύτερα ποια θα είναι τα περιβαλλοντικά αποτελέσματα αυτών των αριθμητικών στοιχείων. Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια πρόσθετα σημεία που νομίζω είναι πολύ σημαντικά. Επίσης, θα ήταν σημαντικό να έχουμε μια γραμμή στο προπολογισμού, έτσι, ώστε ο κάθε βουλευτής να μπορεί να έχει μια επιπλέον βοήθεια για να μπορέσει να εξετάσει και τα αριθμητικά στοιχεία. Τα ταξιδιωτικά οι ταξιδιωτικές δαπάνες ε, των βουλευτών αναφέρθηκαν. Νομίζω ότι είναι δύσκολο να καταλάβουμε γιατί αυξάνονται, νομιώνονται ο αριθμός των βουλευτών και Γενικά οι πράσινοι, και πρέπει να το επαναλάβουμε, λένε ότι το επίδομα γενικών δαπανών χρειάζεται πιο σαφείς κανόνες, θα θέλαμε να μειωθεί και νομίζουμε ότι θα ήταν καλύτερο να έχουμε ξεκάθαρους κανόνες όπως έχει αποφασιστεί από αυτό το Κοινοβούλιο για το συγκεκριμένο επίδομα. Αν ε, δούμε ε, τώρα ε, τις άλλες δαπάνες για το λοιπό προσωπικό είναι πολύ υψηλές αν το συσχετίσουμε με τον αριθμό των ε, βουλευτών και αν δούμε και τι γίνεται με την χρηματοδότηση για τις πολιτικές ομάδες, την ασφάλεια, βλέπουμε αυξήσεις σε όλα αυτά. Και αν τα αντιστοιχίσουμε αυτό στον αριθμό των βουλευτών, έχουμε μαζικές αυξήσεις. Κάτι ακόμα για το οποίο δεν είμαι βέβαιο είναι οι δαπάνε για γενικέ λειτουργίες. Αν δούμε τι αποστολέ των ε, υπαλλήλων έχουμε και πάλι αύξηση εκεί 3,3% στο κόστος και αν ε, το διαιρέσουμε να βουλευτεί έχουμε αύξηση κατά 24% αυτό γιατί ταξιδεύουμε περισσότερο ή γιατί το κόστος ε, του ταξιδίου γενικά αυξάνεται και επίσης εκεί θα θέλαμε μια ανάλυση για τις επιπτώσεις σε ό,τι αφορά τις εκπομπές του εξωτερικού του άνθρακα. Αν δούμε τα κέντρα επισκεπτών, ε, ίσως ε, εγώ ως ε, φιλοευρωπαίος και φεντεραλιστής, εγώ γενικά είμαι υπέρ ε, του να παρουσιάζουμε τη δουλειά μας στο κοινό, αλλά να ρωτιέμαι, έχουμε κάποια αριθμητικά στοιχεία για τα αποτελέσματα του Europe Experience μέχρι τώρα και ο αριθμός ε, των επισκεπτών μπορεί να αξιολογηθεί, δηλαδή υπάρχει κάποιος ε, τρόπος ε, που μας βοηθά να διαδώσουμε τις ιδέες του Κοινοβουλίου ή θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα σε άλλα μέσα, παραδείγματος χάρη στο να έχουμε υλικά κτίρια ή κάποια άλλα μέσα. Νομίζω ότι θα πρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα τον προπολογισμό αναγραμμή, προκειμένου να μπορέσουμε να υπερασπίσουμε, να δώσουμε αυξημένο προπολογισμό και στην πατρίδα μας. Ιδίω ε, αν δεν θέλετε κάποιοι να κάθονται εδώ και να μην έχουν καταλάβει ακριβώς τι γίνεται. Ευχαριστώ κύριο Τσόντσα. Ευχαριστώ. Για τη δική μας πολιτική ομάδα. Εμείς πάντοτε θέλουμε να κάνουμε εξοικονόμηση πόρων. Όμως ε, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνεται εξοικονόμηση πόρων πάση θυσία. Εμείς ε, θα θέλαμε να συγκρίνουμε το μέγεθος του προπολογισμού με την ποιότητα των διοικητικών υπηρεσιών. Χρειάζεται μεγάλος επαγγελματισμό στον τομέα της διοίκησης και αν χρειάζεται περαιτέρω κονδύλια να μας το πείτε. Μιλάμε σήμερα για αυτά τα 89, για αυτές τις 89 θέσεις της ε, Πασαρέλας, δεν είμαστε κατά. Θα πρέπει να προωθήσουμε τις δράσεις που αιτιολογούνται. Εγώ πρέπει να πω ότι φοβάμαι κάπως αυτό το πρασίνισμα του προπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς τι κρύβεται πίσω από αυτό τον όρο. Είχαμε μία επίσκεψη πριν δύο εβδομάδες ε, και είδαμε τα κτίρια και είδαμε ότι υπήρχαν ε, πολλοί σωλήνες, θέρμανσης ε, λοιπά ε, που δεν λειτουργούν ορθά. Δεν ξέρω αν προβλέπονται νέα κονδύλια για αυτές τις εγκαταστάσεις ή όχι. Μιλάμε για το πρασίνισμα του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πώς ακριβώς ε, θέλουμε να καταναλώνουμε την ενέργεια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Ποιε πηγέ ενέργεια θέλουμε να χρησιμοποιούμε. Θα πρέπει επίση να δούμε τη λειτουργία των κτηρίων. Μπορούμε να κάνουμε κάτι συγκεκριμένο ή απλώ ε, θα μιλάμε στη θεωρία. Μπορείτε να μα δώσετε κάποιε λεπτομέρειε σχετικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριο Όλμπριχτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και έχω τρει παρατηρήσει και μία ερώτηση να κάνω στο τέλο. Πρώτη παρατηρήση, ότι ακούγοντα του συναδέλφου, καθίσατε σαφές ότι χρειαζόμαστε ένα πολύ απλό μήνυμα Ποιε είναι οι άμεσε και άμεσε επιπτώσει για το Κοινοβούλιο του Brexit. Μπορεί να μα ε, το θέσουν το ερώτημα αυτό και οι πολίτε, λοιπόν. Εξοικονομούμε χρήματα ή όχι. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά υπάρχουν ε, τα έξοδα τα οποία δεν μπορούμε να περικόψουμε σε ό,τι αφορά τα κτίρια, αλλά θα θέλαμε αυτή την πολύ απλή πληροφορία συνοπτικά. Δεύτερο στοιχείο ως προσωπική παρατηρήση, αν θέλετε, δύο προσωπικές παρατηρήσεις ακόμα συζητάμε τι ανάγκη υπάρχει να διοργανώνονται όλα στο Στρασβούργο. Εκτό από την Ολομέλεια, έχουμε όλο και πιο πολλέ συναντήσει στο Στρασβούργο, όλο και πιο πολλέ αντιπροσωπείε, όλο και πιο πολλέ συναντήσει επιτροπών. Δεν έχουμε τελικά χρόνο να λειτουργήσουμε και να εργαστούμε κανονικά στο Στρασβούργο. Ποιο είναι το κόστο λοιπόν των εργασιών αυτών των επιπρόσθετων στο Στρασβούργο. Αυτό θεωρώ ότι πρέπει να το επιλύσουμε στο μέλλον. Τρίτη παρατήρηση, πολύ προσωπική κάτι ενδεχομένως να μου διαφεύγει, κύριε Γενική Γραμματέα, αλλά ο κορονοϊός. Αυτό το θέμα των ε, χεριών, ε, των βρώμικων χεριών. Ε, τι θα γίνει, δεν μπορούμε να πλένουμε τα χέρια μας στο κοινοβούλιο. Έχουμε κρύο νερό και έρχεται κόσμος, εκατοντάδες, χιλιάδες άνθρωποι σειραίουν εδώ στο κοινοβούλιο. Πώ είναι δυνατόν στο κέντρο τη Ευρώπη να μην έχουμε στο νερό, εν πάση περιπτώσει. Καταλαβαίνω το πρόβλημα που δημιουργείται με τα βακτήρια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κάπως να το επιλύσουμε το θέμα, αυτό το θέμα αυτό, γιατί είναι γελίο. Και τώρα η ερώτησή μου. Το 2021 είναι το πρώτο έτος τη νέα της νέας Και πλέον είμαστε υπό το καθεστώς των νέων υποχρεώσεων του κυρίου Μισελ. Ένα από τα βασικά στοιχεία είναι και πάλι η μείωση του διοικητικού κόστους, ακόμα και σε σχέση με την φιλανδική πρόταση. Τι συνέπειες θα έχει αυτή το, για το Κοινοβούλιο. Μία πρώτη αντίδραση. Καταλαβαίνω ότι πολιτικά δεν είναι πολύ απλά τα πράγματα να κάνετε κάποιε προκαταρτικέ δηλώσει, αλλά θέλουμε να ξέρουμε ω Κοινοβούλιο. Εμεί ω βουλευτέ λέμε όχι, γιατί θεωρώ ότι η μείωση των διοικητικών εξόδων τελικά θα καταλήξει να είναι επικίνδυνη για την σωστή λειτουργία τη διοίκηση. Αυτή είναι η ερώτηση που έχω να κάνω και θα ήθελα μια πρώτη αντίδραση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ο κύριο Στέφαν Ευχαριστώ. Να σας ευχαριστήσω και για την παρουσίασή σας και νομίζω ότι πέρα από αυτά που είπατε, τα οποία τα συνοψίσατε εξαιρετικά, συνάδελφε, έχουμε και άλλο ένα ερώτημα. Το ερώτημα λοιπόν αυτό είναι, θα πολεμήσουμε αυτή τη θητεία για να εξηγήσουμε στους πολίτες τι είναι το Κοινοβούλιο και γιατί θα πρέπει να συμμετέχουν και να ψηφίσουν ή θα κάνουμε πίσω και θα τηρήσουμε υπερσυντηρητική στάση για να δείξουμε ε, αυτοσυγκράτηση. Εδώ λοιπόν ε, έχω να πω το εξή. Το πρόγραμμα το οποίο εφήρμοσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στι προηγούμενε εκλογέ, this time I'm voting, αυτή τη φορά θα ψηφίσω, ήταν πολύ επιτυχέ. Έστειλε πολλά σωστά μηνύματα, γιατί προηγουμένω οι νέοι δεν συμμετείχαν ιδιαίτερα στι εκλογέ. Αυτή τη φορά ήρθαν και ψήφισαν. Έχουμε λοιπόν εκατοντάδες ε, χιλιάδες ε, νέους που περιμένουν μια ηγεσία για το τι θα ακολουθήσει, τι μελεγενέστε. Έχουμε λοιπόν ε, την επιλογή να περιμένουμε μέχρι το 2024 ή να έχουμε μία συνεχή δραστηριοποίηση με τους ανθρώπους αυτούς, τους οποίους έχουμε στις βάσεις δεδομένων μας. Και θα μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους. Να συγχαρώ λοιπόν ε, την ηγεσία του Γενικού Γραμματέα για το This Time I'm Voting, το πρόγραμμα αυτό, ε, είχε μεγάλη επιτυχία. Ένα άλλο καλό πρόγραμμα και έργο, το οποίο το χρησιμοποιούμε κάθε μέρα από όλες τις πολιτικές ομάδες, είναι το EPRS, το οποίο έχει καταστεί το πραγματικό συνεδριακό κέντρο ερευνών. Πριν από δύο θητείες, αν δεν κάνω λάθος, δημιουργήθηκε. Αποτέλεσε ένα πολύ επιτυχές όραμα και χαίρομαι που υπάρχει. Και αν σωστά βλέπω από τα αριθμητικά στοιχεία, αυξάνεται και ο προπολογισμό τους, γιατί αυτό πραγματικά εξοικονομεί δαπάνε για τα θεσμικά όργανα. η Ιδάλω όλα τα κράτη-μέλη θα είχαν ζητήσει μεμονωμένα τέτοιε έρευνε αντί να υπάρχει αυτή η κοινή ομάδα εμπειρογνωμόνων. Και τρίτον, όπως είπε και ο κύριος Σαστέλ, το γραφείο στην να αποτελεί ένα καλό παράδειγμα. Δεν μπορεί να υπάρχει δυσπιστία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Υπηρεσίας εξωτερική δράση. Δεν μπορεί να συνεχίσει ο κόσμος να φεύγει με ιδιωτικέ θεωρήσεις ταξιδίου. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να ασκήσουμε πιέσεις μέχρι να πετύχουμε το αποτέλεσμα για τους βοηθούς των ε, βουλευτών. Η διαφορά μόνο μεταξύ 2020-2021. Νομίζω ότι ήταν στατιστικό όμω το θέμα τη διαφορά αυτό το 3,5%. Είναι θέμα πληθωριστική αντιστάθμισης. Και νομίζω ότι υπάρχει συνήθω θέμα διαμαρρύθμιση και θα ήθελα να με διορθώσετε να κάνω λάθο για τα μίνι τις μίνι και τις ε, κινητές αυτές βουλές αυτή την εμπειρία. Θα ήθελα να έχουμε και πιο πολλές χώρες ε, από την Ανατολική Ευρώπη. Καλό και το Ελτσένκι, είδα και τη Λουμπλιάνα, αλλά πού είναι το Βουκουρέστι, για παράδειγμα. Εξακολουθούμε να μην έχουμε καμία υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί. Και αυτό ενδεχομένω να μας γλιτώσει και χρήματα, γιατί δεν χρειάζεται να στέλνουμε όλους τους πολίτες στις Βρυξέλλες ε, για να επισκεφτούν τους υπέροχους ε, χώρους εργασίας μας μπορούν να του επικεφτούν και εκεί. Τέλο, ασφάλεια. Το είπε ο εισηγητή ο κ. Περέρα. Εγώ θα ήθελα και άλλα μέτρα και μέσα και εργαλεία για εξοικονόμηση πόρων. Speech to text, για παράδειγμα, λογισμικό μετατροπή σε, σε γραπτό λόγο. Αυτό θα σήμαινε μεγάλη εξοικονόμηση κόστου επίση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Χόλμαϊρ. Καταρχάς, να σας καλωσορίσω και την ερώτησή μου την έκανε ο Γιάνν. Θα ήθελα να πω και εγώ για τον Brexit το εξή. Θα ήθελα να ξέρω τι γίνεται με τις συντάξεις των Βρετανών Ευρωβουλευτών. Πώς προβλέπετε το θέμα αυτό. Προσθέσατε και αυτή την ερώτηση, γιατί θα, ξέραμε, θα θέλαμε να ξέρουμε πώς διαμορφώνεται το θέμα των εσόδων-εξόδων σε ό,τι αφορά τον Brexit. Επίσης, κάτι άλλο που με ενδιαφέρει. Για το κτίριο Κόλ. Για την ενημέρωση των υποδομών και των συστημάτων ασφάλειας. Ερωτηματικό εδώ. Ε, επίσης, ε, το κτίριο ΠΑΚ. Ε, να να δούμε τι φταίει λέει η κυρία Χόλμαϊερ. Μήπως να βάλει τα ακουστικά κάτω από το έντρανο. Για το Poland Ring Το κτίριο αυτό. Το λέω αρκετά προσεκτικά. Υπάρχουν ε, διάφορα μόνιμα ερωτήματα. Μέχρι πότε για το κτίριο αυτό θα λαμβάνονται αποφάσεις. Πότε θα ληφθούν οι τελικέ αποφάσει, γιατί αυτό αποτελεί σημαντική επιβάρυνση για τον προπολογισμό, ό,τι και να αποφασίσουμε να κάνουμε. Μιλάμε για μεγάλα ποσά. Και αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει. Και επίσης έχουμε ήδη την εκστρατεία για την ενημέρωση για τις ευρωεκλογέ του 2024, που περιλαμβάνει ήδη τι προβλέπεται για το 2021 και για μόνιμη εκστρατεία ενημέρωσης. Και εδώ θα ήθελα πιο πολλές πληροφορίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Κέλλερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι το δικό μου θέμα αυτό με αφορά και γι' αυτό θα ήθελα να εστιάσω το ενδιαφέρον μου στο κτηριακό. Με τους συναδέλφους, τους σκιώδεις εισηγητές, έχουμε κάνει επισκέψεις σε κτίρια και έχουμε μία βασική ιδέα της τακτικής συντήρησης δεν μιλούμε για ειδικέ εργασίες, για δικές εργασίες. Μιλούμε για ένα ποσοστό που είναι κατά το 2 ή 3% του συνόλου της αξίας του κτηρίου. Αυτό θα μας φαίνεται, μας χρήσιμο. Τώρα, βαριές εργασίες είναι η μόνωση, η θέρμανση, η επισκευή της στέγης. Υπάρχει τέτοια γραμμή στον προϋπολογισμό. Αυτό καταρχάς. Κατά δεύτερο, για το Europa Experience. Θα ήθελα να μιλήσω για το ενδιαφέρον που έχει αυτός ο μηχανισμός. Και θα ήθελα να παρακαλέσω να γίνουν αυτές οι δαπάνες οι οποίες πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση, προς την κατεύθυνση της ε, βελτίωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έχουμε και τα νέα κρατημέλη. Τώρα το Κοινοβούλιο με την νέα θητεία και την προσχώρηση των νέων μελών έχει φτάσει πια στην εφηβεία του. Είδα την παρουσίαση με πολλά επιχειρήματα στην έκθεσή σας, αλλά δεν βρήκα στο, τη γραμμή του προϋπολογισμού στην συθνετική απεικόνηση ε, του κεφαλαίου, κεφαλαίου 20.7. Παρ' όλα αυτά τα ποσά είναι σημαντικά. Τρίτο ερώτημα για το κτίριο Σπινέλη, Αλτιέρο Σπινέλη, το οποίο και εμείς επισκεφθήκαμε και μελετήσαμε σε βάθος. Ευχαριστώ τον μιλό. Είδαμε τους ηλεκτρικούς μετασχηματιστές ε, και τα μπόιλερ που θα πρέπει να αντικατασταθούν. Τους καυστήρες δηλαδή. Ε, δεν βλέπω αντίστοιχες γραμμές στον προϋπολογισμό για το Σπινέλι. και είναι σημαντικά αυτά. Βλέπω τα τις αίθουσες των εστιατορίων, αλλά όχι τα πιο τεχνικά ζητήματα να μην υπάρχουν σε γραμμή προεπολισμού. Η Μόνικα Χολμάγερ γνωρίζει πολύ καλά το θέμα αυτό. Ε, θα ήθελα να σας πω ότι πρέπει να δουλέψουμε γρήγορα τώρα. Και με εκπλήσει το γεγονό ότι βλέπουμε να εμφανίζονται 10 εκατομμύρια ευρώ, 10,3 εκατομμύρια ευρώ για το κτίριο Πόλαν Ρι Σπακ, χωρίς να έχουμε καμία ιδιαίτερη πληροφόρηση και ενημέρωση. Εγώ εισηγήτρια και δεν έχω ιδέα για το τι συμβαίνει και γιατί χρειάζεται να γίνουν δαπάνες ύψους 10,3 εκατομμυρίων ευρώ για το κτίριο Πολ Ανρί Σπακ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η κυρία Γκουάρδια Θαμπάλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολλές ερωτήσεις έχουν τεθεί. Δεν θέλω να επαναλάβω τα ίδια. Θα θίξω δύο ζητήματα που άπτονται τρόπον την άτο προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρώτον, τις συνθήκες εργασίας των ε, ε, εργαζομένων στις υπηρεσίες καθαρισμού. Κατά κύριο λόγο πρόκειται για γυναίκες. Έχει γίνει πάρα πολλές φορές συζήτηση για αυτό το θέμα. Οι υπηρεσίες του Κοινοβουλίου μας λένε ότι τηρούν τον νόμο. Αυτό τους έλειπε κιόλα, αλλά προσθέτω εγώ, αλλά είναι μία είναι οι συνθήκες που δίδονται στις καθαρίστριες από την εταιρεία που τις επινοικιάζει ε, οι συνθήκες που, για τις οποίες αγω, εμείς αγωνιζόμαστε για ε, αξιοπρεπή εργασία. Εάν ε, ζητούμε αξιοπρεπείς συνθήκε εργασίας έξω στην αγορά στις χώρες μέλη, ε, τότε να ξεκινήσουμε μετά του οίκου μας και να προσφέρουμε αξιοπρεπείς συνθήκε εργασίας στους εργαζομένους μας, ε, στις εργαζόμενες στην υπηρεσία καθαρισμού. Για τους υπότροφους μας πήρε πέντε χρόνια να, να κερδίσουμε αυτή τη ε, μάχη. Από εκεί και πέρα υπάρχουν αποφάσεις επιτροπής μας και υπάρχει ε, διαφορά αρμοδιοτήτων με τις αποφάσεις του Προεδρείου. Συχνά υπάρχουν αποφάσεις από το Προεδρείο που έρχονται στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και δεν μπορούμε να απορρίψουμε καλύψουμε διότι έχουν ήδη εγκριθεί, αλλά πρέπει να βρούμε χρηματοδότηση μέσα στον προπολογισμό. Και αυτές οι διαπραγματεύσεις που πρέπει να κάνουμε με το Προεδρείο είναι κάπως επίπονες και μας περιπλέκουν ενίοτε τη ζωή διότι έχουμε και το στόχο να μην ξεπεράσουμε την αύξηση του προπολισμού κατά χ ποσοστιαίε μονάδες και το καθεξής. Αλλά μπορεί να συμβεί και το αντίθετο και γι' αυτό το είπα αυτό ω εισαγωγική παρατήρηση. Τι εννοώ, σε πάρα πολλές ολομέλειες πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει υπερψηφίσει συγκεκριμένε προτάσει, οι οποίε τελικά μπλοκαρίστηκαν για διάφορου λόγου. Θα σας δώσω δύο παραδείγματα. Στο τέλος της προηγούμενης θητείας ζητήσαμε οι βοηθοί να τους επιστρέφονται τα έξοδά τους στο ίδιο επίπεδο με τους ε, δημοσίους λειτουργούς, με τους δημοσίους υπαλλήλους, τους μόνιμους όταν πάνε σε αποστολή και κατά κύριο λόγο φυσικά στο Στρασβούργο. Να μην παίρνουν λιγότερα δηλαδή ως έξοδα αποζημίωσης ταξιδίου και ούτε καθεξής. Το Κοινοβούλιο το ενέκρινε αυτό και παρέλυσε το ζήτημα. Δεν έγινε τίποτα. Ζητήσαμε το Προεδρείο να μελετήσει τεχνικές δυνατότητες ώστε ένας βουλευτής ή μια βουλεύτρια που έχουν άδεια μητρότητας ή πατρότητας να μπορεί να ψηφίσει διαδικτυακά γιατί δεν μπορεί να πάει στην Ολομέλεια για το χύψη λόγο. Όπως επίσης ε, για, ε, το ίδιο να ισχύσει και για βουλευτές που μπορεί να πάσουν από κάποια νόσο, μακροχρόνια και το καθεξής και δεν μπορούν να μεταβούν στην Ολομέλεια, να μπορούν να ψηφίσουν ηλεκτρονικά. Εγκρίθηκε αυτό, αλλά παρέλυσε, δεν προχώρησε. Δηλαδή, ε, το, πρόεδρο, αν το Προεδρείο λαμβάνει αποφάσει τι οποίε εμεί μετά πρέπει να κόψουμε το λαιμό μα, να βρούμε τρόπο να τι εφαρμόσουμε και πόρου και ε, γραμμέ στον προπολογισμό, τότε θα θέλαμε και το Προεδρείο από την πλευρά του τι δικέ μα αυτέ αποφάσει που έχουμε ψηφίσει να τι προχωρήσει και να μην τι αφήσει ω θέματα ε, σε τέλμα. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο στον κύριο Βέλε για να απαντήσει. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, και θα προσπαθήσω στο βαθμό του δυνατού να απαντήσω όλε τι ερωτήσει αυτέ. Καταρχά, να ευχαριστήσω τον εισηγητή και για την καλή συνεργασία μεταξύ άλλων. Η πρώτη ερώτηση ήταν τι γίνεται με το περιβαλλοντικό καθεστώς σε ό,τι αφορά τα κτίρια τα μας. Το θετικό είναι το εξή. Στα καινούργια κτίρια και κυρίως στο κτίριο Μάρτενς, έχουμε πραγματικά εξαιρετικό καθεστώς. Ε, είναι το πιο υψηλό καθεστώ, τα πιο υψηλά πρότυπα ε, που υπάρχουν. Υποδειγματικό κτίριο. Η... Ο παιδικό σταθμό Weinberg, ο οποίο ανακαινίζεται, θα είναι παθητικό κτίριο. Στο κτίριο Adenauer, το οποίο έχει ολοκληρωθεί κατά 70%, χρησιμοποιούμε ε, γεωθερμική θέρμανση και με κλιματισμούς. Χρησιμοποιείται δηλαδή ε, γεωθερμική ενέργεια σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα πρότυπα και προσπαθούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τεχνικές εγκαταστάσεις οι οποίες από οικολογικής άποψη είναι εξαιρετικέ. Στο ό,τι αφορά το θέμα ε, των μεταφορών. Τα τελευταία χρόνια έχουμε αλλάξει σημαντικά τον τρόπο μεταφορά των υπαλλήλων μας. Χρησιμοποιούμε πλέον τρένα θαλή σε ό,τι αφορά τη μεταφορά στο Στρασβούργο και δεν βασιζόμαστε πλέον δηλαδή στις ε, μεταφορές ε, με γιοδαχή. Είναι μεγάλο, μεγάλη πρόοδος αυτή και έτσι χρησιμοποιούμε ηλεκτρικά δίκτυα. Έχουμε 111 μάλλον θέσεις στάθμευσης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, για ανεφοδιασμό ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Και το Προεδρείο αποφάσισε το 2019 στη φάση προσαρμογής να μπορεί να έχει κανείς ένα εποχικό συντηρίο και για έξι μήνες για να μπορεί ως τώρα κάθε υπάλληλο ε, είχε δικαίωμα να έχει χώρου στάθμευσης. Εμείς ε, λοιπόν προσφέρουμε τώρα αυτή την ευκαιρία εάν οι υπάλληλοι αποφύγουν και δεν χρησιμοποιήσουν αυτό το δικαίωμα. Θεωρούμε ότι είναι ένα καλό σύστημα για να κάνουμε μετακίνηση από το προσωπικό τρόπο μεταφοράς ε, στις μαζικές συγκοινωνίες. Έχουμε αντικαταστήσει λοιπόν ε, και διάφορα γεωταχή με υπηρεσιακά οχήματα. Και εδώ λοιπόν προωθούμε την πιο φιλική προς το περιβάλλον μεταφορά. Στις Βρυξέλλες λοιπόν επίσης προτείναμε για να αποφύγουμε περιττές μεταφορές μεταξύ των δοσμικών οργάνων, να υπάρχει σύνδεση μεταξύ. Εμείς παρουσιάζουμε το σχέδιο και ο Δήμος θα το αμα, ο σχέδιο, να υπάρχει υποδηλατά δρόμος για τη σύνδεση των θεσμικών οργάνων στις Βρυξέλλες. Το ερώτημα τώρα για την κτηριακή πολιτική 2029 πρόκειται για μια κτηριακή πολιτική η οποία ψηφίστηκε ήδη το προηγούμενο Προεδρείο για μια μακροπρόθεσμη λοιπόν στρατηγική για τα κτηρία. Το Κοινοβούλιο αποφάσισε ότι πλέον έχουμε επαρκή γραφεία εδώ στις Βρυξέλλες ιδιαίτερα αλλά και στο Στρασβούργο με τα μέτρα που επλέον λήφθησαν. Και έτσι λοιπόν θα πρέπει να τεθούν ε, νέε προτεραιότητε. Η εμπειρία τη Ευρώπη για του πολίτε, για την ενημέρωση των πολιτών, η δυνατότητα διεξαγωγή ε, τριμερών διαλόγων ε, σε κατάλληλε καταστάσει και η ανακαίνιση. Η ανακαίνιση είναι σημαντικό σκέλο, να σα επισημάνω. Θεωρούμε ότι τη στιγμή που ένα κτίριο έχει κλείσει 25-30 χρόνια χρήση, χρειάζεται τουλάχιστον ενεργειακό πώ να γίνει η εξυγίανση και ως ε, ε, νομοθέτης ε, αποφασίσαμε και υποχρεώσαμε και τους ιδιωτικούς ιδιοκτήτες να αφιερώνουν 3% σε ανακαίνιση των Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι σε 33 χρόνια θα πρέπει να έχει ανακαινιστεί το σύνολο των κτηρίων. Σε ό,τι αφορά το αυτό που αναφέρατε, τη συγκεντρώση αυτή. Νομίζω ότι τα τελευταία δύο χρόνια είχαμε 30 δις ευρώ, δηλαδή δαπανήθηκε 98,5% του προπολογισμού. Είναι υψηλό ποσοστό απορρόφηση του προπολογισμού, 150 80 εκατομμύρια ευρώ την πέρσι. Εδώ θεωρούμε λοιπόν ότι έχει μειωθεί αυτό το όραμα Αυτό που είναι θετικό είναι ότι αυτό σημαίνει εξοικονόμηση τόκων. Εδώ θεωρούμε ότι τα κτίρια στο Λουξεμβούργο αμα, γλιτώσαμε 100 εκατομμύρια ευρώ γιατί δεν ε, αμ, καταβάλαμε τους τόκους. Θεωρώ λοιπόν ότι ήταν ε, σκόπιμο αυτό το μέτρο συγκέντρωσης των εξόδων σε ό,τι αφορά και το όφελος το οποίο είχε ο Ευρωπαίος προλογούμενος. Σε ό,τι αφορά τη στρατηγική μας, το Προεδρείο δήλωσε ότι ήθελε υψηλότερο επίπεδο φιλοδοξία και έκανε μια πρόταση λοιπόν το Προεδρείο σε ό,τι αφορά όλους του στόχους για το Πράσινο Κοινοβούλιο. Είτε να συνεχιστούν αυτοί οι στόχοι, είτε να διαμορφωθούν με, σε πιο φιλόδοξο επίπεδο ή και τα δύο. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά το διοξείδιο του άνθρακα, θέλουμε μείωση 40% μέχρι το 2030. Το Προεδρείο τώρα αποφάσισε 40% μέχρι το 2024. Σε ό,τι αφορά την μεταφορά των ατόμων, 20% ε, μέχρι το 2030, τώρα αποφασίσαμε 30% μέχρι το 2024. Αυτό σημαίνει δηλαδή στο ίμιση του χρονικού διαστήματος που προβλέπονταν αρχικά. Σε ό,τι αφορά τη μείωση 15% μέχρι το 2025, τώρα έχουμε το 25% μείωση μέχρι το 2024. Ανεώσιμες πηγέ ενέργεια. 10% μέχρι το 2025, τώρα είμαστε στο 25% μέχρι το 2024. Η ηλεκτρική κατανάλωση, στόχος μείωσης 20% μέχρι το 2024 σε ό,τι αφορά την κατανάλωση χαρτιού. Παλιό στόχο 15% μέχρι το 2025. Τώρα είμαστε στο 50% μέχρι το 2024. Νέο στόχο. Κατανάλωση νερού 2%. 15% και ούτω καθεξή μπορώ να σα δώσω πολλά στοιχεία τέτοια να σα ενδιαφέρουν. Να σας πω λοιπόν ότι το νέο Προεδρείο τους στόχου για το περιβάλλον τους ε, μετατόπισε χρονικά σε πιο έγκυρο χρονικό σημείο ή αύξησε το επίπεδο φιλοδοξία. και αυτά θα πρέπει να αποφασιστούν ως ε, μεμονωμένα μέσα και μέτρα για να μπορέσουν να υπάρχουν ρεαλιστικοί στόχοι. Επίσης, μιλήσατε για την εξωτερική παρουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εδώ και 10 χρόνια έχουμε γραφείο στην Ουάσιγκτον και θεωρώ ότι λειτουργεί πάρα πολύ καλό. Πριν από 10 χρόνια Μα ρωτούσαν στην Ουάσιγκτον και μα έλεγαν «Α, μάλιστα, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ήρθατε». Όχι, πλέον κομμάτια αυτά. Ούτε στο Κογκρέσο, ούτε πουθενά αλλού. Έχουμε αποστείλει και πάνω από 200 βουλευτέ ε, στο Κογκρέσο. Και έχουμε πετύχει λοιπόν διαφορέ τέτοιες, ε, τέτοια επιτεύγματα. Αυτό δεν είναι η κλασική ε, εξωτερική πολιτική όπως έχει υπόψη της υπηρεσία εξωτερικής δράσεις. Για παράδειγμα, στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών μπορεί κανείς να συμμετέχει σε συνεδριάσεις ή, για παράδειγμα, πολιτική δική μας από τον τομέα μεταφορών, των γεωργικών. Πρόκειται για τέτοια συγκεκριμένη συνεργασία και γι' αυτό, λοιπόν, θεωρώ ότι είναι και νόμιμη η παρουσία των Ευρωβουλευτών. Και το ίδιο ισχύει και για το Λονδίνο. Θα συνεχίσουμε να έχουμε παρουσία στο Λονδίνο, αποφασίστηκε. Έχουμε 2,7 ε, εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες στην, ε, στο Λονδίνο. Δεν μπορούμε λοιπόν να συμπεριφερθούμε πλέον μετά το Brexit στο Λονδίνο, λες και πρόκειται για ένα οποιοδήποτε τρίτο κράτος. Θα πρέπει να ασχοληθούμε με αυτούς που ζουν εκεί και έχουν σημαντικά προβλήματα και σημαντικά συμφέροντα στην περιοχή. Το Προεδρείο επίσης πέραν τούτο αποφάσισε να έχει παρουσία στις ε, πολυμερείς οργανισμούς με εκπρόσωπο των ΟΗΕ, των ΑΣΕΑΝ, στην Αφρικανική Ένωση και νομίζω ότι σε τέτοιους καιρούς όπου απειλείται η πολυμέρεια είναι σημαντικό μέτρο αυτό. Επίσης, ε, μας είπατε τι γίνεται με τις ε, υλοποίησεις των αποφάσεων Χάσελμορ. Έχουμε εδώ μια επισκόπηση σε σχέση με το τι έχει υλοποιηθεί από το σχέδιο δράση. Να σας πω ότι δεν υπάρχει τίποτε με κόκκινο χρώμα το οποίο δεν έχει υλοποιηθεί καθόλου. Τα πιο πολλά είναι στο 75%-80% πράσινα. Υπάρχουν και κάποιοι τομεί με κίτρινο που χρειάζονται περαιτέρω εργασία. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια νέα φάση όπου η κάθε απόφαση που έχει ληφθεί θα πρέπει να αποδέξει την αξία της στην πράξη. Έχουμε ένα νέο σύστημα λοιπόν στη νέα θετία και το Προεδρείο καλά θα κάνει σε κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα 18 μήνες ενδεχομένως να εξετάσει κατά πόσον ε, επιτεύχθησαν οι στόχοι που είχαν τεθεί για κάθε μέτρο ή... Όχι. Προκειμένου ανάλογα να προσαρμοστούν και τα μέτρα. Η ε, κυρία Βίντσικ έθεσε το εξής ερώτημα. Τι γίνεται με την προεκλογική εκστρατεία. Κατά τη διάρκεια των ευρωεκλογών είχαμε πολύ θετικέ εμπειρίες με μια διαφορετική παρουσία σε ό,τι αφορά τους πολίτες σε πολλά επίπεδα. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τα εξωτερικά γραφεία. Είχαμε εμπειρογνώμονες και για τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, οι οποίοι ενίσχυσαν ε, το έργο μας ό,τι αφορά τη δημοσιότητα. Επίσης, δραστηριοποιηθήκαμε και σε κεντρικό επίπεδο με διαφορετικό τρόπο, για παράδειγμα το είπε ο Στέφαν Χούτα. Ε, είχαμε την καμπάνια What Europe Does For Me. Είχαμε 300.000 ε, πολίτες οι οποίοι δικτυώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δήλωσαν ότι θέλουν να κάνουν εκστρατεία. Είναι σημαντικό αυτοί οι 300.000 ε, πολίτες να μην περιμένουν 4-5 χρόνια μέχρι ότου ξανασυνεργαστούν με το Κοινοβούλιο, να αντιτρήσουμε την επαφή με τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι φροντίζουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θέλουν να εργαστούν για την Ευρώπη. Και επίσης κάτι πολύ συγκεκριμένο για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην διαπραγματεύονται μόνο οι βουλευτέ να παρακολουθείτε από το κοινό η διαδικασία αυτή. Αυτό και στην διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Δεν μπορούμε δηλαδή να πάμε στις εκλογές μία φορά και τελείωσε. Χρειάζεται μία διαρκής παρουσία. Ρωτήσατε επίσης για την ευρωπαϊκή αυτή εμπειρία, για τα κινητά αυτά κοινοβούλια. Για να σας δώσω ένα πρακτικό παράδειγμα. Πριν από κάποιο καιρό, πριν από κάποιες μήνες μάλλον, για πρώτη φορά αυτή η ευρωπαϊκή εμπειρία ξεκίνησε στο Ελσίνκι, στην καινούργια Εθνική Βιβλιοθήκη στο Ελσίνκι. Πριν ε, είχαμε ένα έτος 3.000 επισκέπτες, τώρα έχουμε 130.000 επισκέπτες. Αυτό σημαίνει ότι αυτό το ευρωπαϊκό, αυτή η ευρωπαϊκή εμπειρία αποτελεί μια ευκαιρία για να περάσουμε σε ένα επίπεδο μαζικής επικοινωνίας, όχι εντελώ εξειδικευμένη παρουσία. Σα το λέω και για το Στρασβούργο. Από τότε που ξεκίνησε έχουμε 460.000 επισκέπτες στο Στρασβούργο και στο Παρλαμεντάριο εδώ στι Βρυξέλλε. 2,5 εκατομμύρια επισκέπτες εδώ λοιπόν έχουμε πραγματικά μία ευκαιρία να έχουμε μαζική επικοινωνία σε μεγάλο εύρο φάσματο σε ό,τι αφορά του επισκέπτε. Γι' αυτό λοιπόν και το Προεδρείο αποφάσισε να είναι γενική αυτή η διάσταση. έχουμε γενικά τέτοια έργα σε όλες τις πρωτεύουσες, όχι μόνο στις ε, Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο. Και στο Ταλίν προγραμματίζεται το επόμενο έργο, 15 Μαρτίου, ξεκινά στο Ταλίν επειδή για τι ανατολικέ χώρες, τι βαλτικέ χώρες, ε, ένα τέτοιο ευρωπαϊκό έργο και ελπίζουμε επενδύουμε μάλλον στις χώρες εκείνες οι οποίες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις σε ό,τι αφορά το σκέλος της επικοινωνίας. σε ό,τι αφορά κάποιες γραμμές του προπολογισμού, ενδεχομένως να υπάρχει κάποια σύγχυση. Γιατί βλέπουμε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά που είχαμε συνηθίσει. Γιατί πρόκειται για αριθμούς οι οποίοι είναι διαιρεμένοι για δύο έτη. Όχι λοιπόν 11, κάτι εκατομμύρια, αλλά 8 εκατομμύρια, γιατί εδώ συμπεριλαμβάνονται περισσότερα από ένα νομοσυνομικά έτη. για το Λουξεμβούργο. Η διαδικασία προκήρυξη διαγωνισμών για δημιουργία καταλόγου αποθεματικού. Χρειαζόμαστε τέτοιο κατάλογο να υπάρχει για ένα έτος ήδη. Ένα έτος πριν να ξεκινήσει η διαδικασία. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα ε, προσληφθούν οι άνθρωποι αυτοί απαραίτητα από 2021 και μετά ενδεχομένω να προσλάβουμε. Για το Brexit τώρα ακούσαμε ένα ερώτημα γιατί δεν υπάρχουν ε, περικοπές ε, σε ό,τι αφορά τις γραμμές του προπολογισμού που έχουν να κάνουν με το προσωπικό και τις μεταφορές. Ο λόγος είναι ότι ο... το έτος που υπολογίστηκε το Brexit ήταν το 2019. Το 2019 λοιπόν είχαμε υπολογίσει ότι θα έχουμε ήδη πιο λίγους βουλευτές ότι θα χάνουν περίπου 600 ε, βουλευτέ, Δεν προέκυψε προφανώ αυτό και γι' αυτό υπάρχουν ε, τόσο μικρές διαφορές. Τα έξοδα και τα πάνες υπολογίζονται επίσης ε, βάσει των μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας. Σε ό,τι αφορά τους βοηθούς, σε κάποιε περιπτώσει οι βουλευτέ δεν εξαντλούν το πόσο που προβλέπετε. Και Θεωρούμε, για παράδειγμα, ότι αυτά τα έξοδα θα γίνουν. Βλέπουμε, για παράδειγμα, ότι πολλοί βουλευτέ θα χρειαστούν τέταρτο βοηθό και βλέπουμε ότι θα είναι πιο μεγάλη η συμμετοχή των πολιτών σε ό,τι αφορά τι και σε άλλε κοινοβουλευτικέ δραστηριότητε. Γι' αυτό θεωρούμε ότι θα χρειαστεί προσαρμογή των δαπανών για την πολιτική για το διοξείδιο του άνθρακα. Σα είπα πόσο πιο φιλοδοξή είναι η στόχη. 43% μέχρι το 2024, όχι μέχρι το 2030 και κυρίως ό,τι αφορά την ε, μετακίνηση. Το ποσό καταποκοπής πάντα είναι θέμα στο Προεδρείο και σίγουρα θα παραμείνει για τα γενικά έξοδα, για τις γενικές δαπάνες. Για την εμπειρία της Ευρώπης Experience ε, Europe ε, σας τα είπα για τις 89 αυτές ε, καινούργιε θέσεις δεν θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερο κόστος, μεγαλύτερες δαπάνες, γιατί θα χρησιμοποιηθούν από υπαλλήλους οι οποίοι θα συνεχίσουν να απασχολούνται από πολιτιστικές ομάδες. Είναι τεχνική η αλλαγή αυτή, δεν σημαίνει επιπλέον κόστος. Και είπατε και για το κόστος των νέων ενεργειακών ε, πηγών. Σας είπατε χρησιμοποιούμε τη γεωθερμική ενέργεια στο Λουξεμβούργο και με τον καλύτερο τεχνικό εξοπλισμό θεωρούμε ότι θα έχουμε καλύτερη αξιοποίηση της ενέργειας. Ο πρόεδρος. Κλάους, βλέπω ότι έχεις πολλές σημειώσεις. Αλλά έχουμε να ξεκινήσουμε και το επόμενο σημείο. Ναι, ναι, ναι. Να απαντήσω όσο μου δίνετε χρόνο. Κύριε Ολμπρέχτ, για το Στρασβούργο και τα επιπλέον, ε, τις επιπλέον Επιπλέον Ο, το κόστος της τριπλής έδρας είναι 100 εκατομμύρια το χρόνο. Το το κρύο νερό. Έχουμε πρόβλημα με το βακτήριο της λεγιονέλας. Το πρόβλημα είναι ότι ε, αν δεν χρησιμοποιούνται τακτικά οι βρύσες μέσα στο νερό, υπάρχει η πιθανότητα να αναπτυχθεί το βακτήριο αυτό και γι' αυτό έχουμε κρύο νερό. Να τα κάνω λίγο τροχάτα τα υπόλοιπα. η κυρία Χόλμαϊρ μίλησε για το Ταμείο Συνταξιοδότησης. Δεν μας ε, αγγίζει άμεσα το θέμα των συντάξεων, αλλά σε ό,τι αφορά το εξωτερικό Ταμείο θα χρειαστούν περαιτέρω εξηγήσει γιατί δεν μου δίνει χρόνο ο πρόεδρο. Για το κτίριο Κόλ. Ναι, μου το επιτρέπετε, μου το επιτρέπετε. Να σα πω λοιπόν τι γίνεται σε ό,τι αφορά τι συντάξει. Εδώ έχουμε ένα σημαντικό έλλειμμα το οποίο οι υπόλοιπε συντάξει δεν περιλαμβάνονται στον προπολογισμό του Κοινοβουλίου. Σε ό,τι αφορά το κτίριο Κόλλα, χρειαζόμαστε ανακαίνιση και γιατί γίνονται και εκεί τριμερεί διάλογοι. Δεν είναι αποδεκτό έτσι όσο έχει. Σε ό,τι αφορά το κτίριο PHS, έχει γίνει μια ε, προκήρυξη διαγωνισμού και στην επόμενη θητεία θέλουμε να ξεκινήσουμε το 2024 περίπου τις εργασίες για την ανακαίνιση. Κυρία Κέλλερ ρωτήσατε για την τήρηση του 3%. Αυτό είναι απαραίτητο. Γι' αυτό υπάρχει μια νέα διεύθυνση η οποία ασχολείται μόνο με το θέμα αυτό σε ό,τι αφορά και την ε, αρχαιότητα των κτηρίων μας. Αλλά αυτό διανέμεται σε διάφορες, ε, σε διάφορες κεφάλαια του προπολογισμού. Αν θέλετε δημερώσω να σας τα εξηγήσω. Ευχαριστώ για το κτίριο ΣΠΑΚ επίση ετέθησε το ερώτημα το τι θα γίνει. Ο κύριος Στέφανο αναφέρθηκε σε αυτό και συμφωνώ και το EPRS και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, η οποία επίσης πρέπει να ανοίξει. Η παλιά αυτή αυστηρή διάκριση μεταξύ των πολιτική, δεν υπάρχει πλέον και το κλίμα και η πολιτική άλλες πολιτικές υπάγονται πλέον στις εσωτερικές πολιτικές. Η κυρία Γκαρδία Ζαμπάλ μίλησε για την κατανομή των εργασιών. Είμαστε σε φάση διαρκούς εποπτείας, κάνουμε προσπάθειες να εγγυηθούμε σωστή λειτουργία των υπηρεσιών μας. Τελευταίο θέμα για το θέμα του Προεδρείου και της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Όντως, εδώ υπάρχουν διαφορετικές τοποθετήσεις και ο καθένας έχει λίγο διαφορετικό ρόλο σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ερώτημα των ε, βοηθών, έχουμε τρία διαφορετικά καθεστώτα για τους βουλευτές, για τους υπαλλήλου και για τους ε, βοηθούς. Ε, γίνεται έντονη συζήτηση στο Προεδρείο για αυτά και το Προεδρείο πλειοψηφικά αποφάσισε τρία διαφορετικά συστήματα να υπάρχουν, αλλά σε ό,τι αφορά τα σχετικά επιδόματα αποφάσισε αναλόγω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και ο Πρόεδρο, για την παρουσία σα και για την παρέμβασή σα. Και τώρα να δώσουμε το λόγο στον Αντιπρόεδρο και κύριο Περέρα. Γιατί έχουμε καθυστερήσει και πρέπει να ξεκινήσουμε και με το επόμενο σημείο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θα είμαι πολύ συντομό. Απλώς δύο καταληκτικά σχόλια. Όπως είπα στην αρχή, σε αυτό το στάδιο, αυτό είναι ο προπολογισμό του Γενικού Γραμματέα, ο οποίος ε, θα υιοθετηθεί από ε, το Προεδρείο στις 9 Μαρτίου και επομένως οι συνεισφορές σας στο στάδιο αυτό είναι πολύ σημαντικές για μας και για τη συζήτηση που θα έχουμε σε επίπεδο Προεδρείου. Τα δύο σχόλια που θέλω να κάνω είναι το εξή. Ε, καταρχήν να πω ότι σημειώνω την αναγκαιότητα να γίνει μία πρόσθετη προσπάθεια για να διαδώσουμε τα όσα κάνουμε και στη διαχείριση του Κοινοβουλίου, ε, γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει κατανοητό ο προπολογισμό. Εμείς βλέπουμε επενδύσεις σε κτίρες συνθήκες εργασίας ε, και σε εξοπλισμό. Αν ε, όμως ε, μάλλον πρέπει να δούμε και την στρατηγική που υπάρχει για τα κτίρια που καταρτίστηκε το 2010 και ανανεώθηκε το 2018 και αυτό σημαίνει εξοικονόμηση πόρων ε, σε σχέση με εναλλακτικά σενάρια ε, για την ανακαίνιση των κτιρίων. Έτσι λοιπόν το θέμα ε, της περιουσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, ουσιαστικά δομήθηκε με έναν τρόπο που αφορούσε και εξοικονόμηση των πόρων. Ε, ένα άλλο θέμα έχει να κάνει με το Πράσινο Κοινοβούλιο. Εγώ βλέπω ότι κάποιες από τις προσπάθειες που γίνονται για να μπορέσουμε παρούντος χάρη να μειώσουμε τις εκπομπές και το τι κάνουν σχέση με τους οδηγού. δεν είναι αυτά απόλυτα γνωστά στους βουλευτές. Πρέπει λοιπόν λοιπόν το Προεδρείο να διαδώσει περισσότερο αυτές τις πληροφορίες, γιατί αν εμείς οι ίδιοι δεν γνωρίζουμε, τότε και έξω πολύ λιγότερο γνωρίζουν το τι κάνουμε. Και κάτι τελευταίο για τον Brexit. Να πω ότι εγώ καταλαβαίνω πολύ καλά το, αν δούμε τις επιπλοκές και τις επιπτώσεις του Brexit σε ό,τι αφορά τη συγκράτηση των πόρων του Κοινοβουλίου, όμως ε, η μεγάλη πρόκληση που θέτει το Brexit είναι πώς ε, θα απαντήσουμε στις επιθέσεις κατά του ευρωπαϊκού σχεδίου, κατά του λαϊκισμού και πώς ε, θα επενδύσουμε στην διάδοση των ευρωπαϊκών αξιών. Και προγράμματα όπως το Europa Experience έχουν απόλυτο νόημα και Μπορούμε λοιπόν να αφιερώσουμε με τον προπολογισμό σε αυτά. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Θα τα συμπεριλάβουμε και στην συζήτηση που θα αφορά αυτή τη δημοσιονομική πρόταση. Μάλιστα, εδώ ολοκληρώνουμε αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ τους ε, προσκεκλημένους για τις ε, παρουσιάσεις τους. Ευχαριστώ και τον ε, κύριο Σαστέλ που δεν θα κάνει καταληκτικές παρατηρήσεις γιατί έχουμε καθυστερήσει και 10 λεπτά και θα περάσουμε στο επόμενο σημείο. Είναι μια κοινή συνάντηση τριών επιτροπών για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.